τυπικό. Το Ευρωπαϊκό, ε, συγγνώμη, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, υπέβαλε διορθώσεις σε τρία κείμενα. Σήμερα με το άρθρο 2.31.4 θα θεωρηθεί ότι ε, ισχύουν αυτές οι διορθώσεις αν δεν έχουν αναγγείλει μέσα σε 24 ώρες διορθώσεις και αντιρρήσεις. Μια πολιτική ομάδα τουλάχιστον 40 βουλευτές. Το κείμενο είναι στον, στο χώρο του Κοινοβουλίου. Τα κείμενα και οι διορθώσεις. Τώρα θα έχουμε τη δήλωση του υποψηφίου για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής